Αγαπητοί συνάδελφοι, με ιδιαίτερη χαρά κηρύσω την έναρξη της έκτακτης αυτής συνεδρίας της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και καλωσορίζω την ύπατη εκπρόσωπο τη Βαρόνη Κάθριν Άστον. Και ε, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που αντικαθιστώ σήμερα τον κύριο Μπρόκ στην Προεδρία. Χρειάστηκε να μείνει στην Γερμανία γιατί έχει μια ανελημμένη υποχρέωση έπρεπε να παραβρεθεί στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Καλσρούης. Απόλυτα δικαιολογημένη η απουσία του. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τη Βαρόνια Άστον για το έργο που έχει επιτελέσει στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, γιατί οι επόμενοι μήνες θα είναι πραγματικά κρίσιμοι για την επιτυχία αυτών των διαπραγματεύσεων και εκτιμούμε ιδιαίτερως όλοι το γεγονός ότι εσεί ε, κυρία Άστον, Δηλώσατε ρητά ότι θα συνεχίσετε τις προσπάθειες και προσωπικά για να εξασφαλίσετε την τήρηση των υποσχέσεων και των όρων που ε, ανέλαβε το Ιράν να τηρήσει. Δυστυχώς όμως το Ιράν δεν είναι το μόνο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Η επιτυχής ε, έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης επίσης είναι κρίσιμη σημασία για την σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Οπότε η συνέχιση του διαλόγου προκειμένου να βρεθεί πολιτική λύση και στη σύγκρουση της Συρίας είναι θεμελιώδη σημασία αν θέλουμε να αποφύγουμε μια καταστροφή όχι μόνο ανθρωπιστικού χαρακτήρα αλλά και πολιτικού και μια διάλυση εθνοτική και θρησκευτική της Συρίας και ε, με ιδιαίτερες συνέπειες για τις γειτονικέ χώρες. Και να ολοκληρώσω με δύο σχόλια. Ε, θα θέλαμε ε, να μάθουμε τι γίνεται με την Ουκρανία επίσης, ε, ποιες είναι οι πολιτικές εξελίξεις ε, για την Ουκρανία, αν υπάρχουν βάσεις για να επιχειρήσουμε μία διαμεσολάβηση και αν είναι δυνατόν να αλλάξουμε την πολιτική πορεία που φαίνεται ότι ακολουθεί ο πρόεδρος Γιαννουκόβιτς. Και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την υπογραφή της συμφωνίας. Και ιδιαίτερα Άλλο σοβαρό θέμα είναι το θέμα της Κεντροαφρικανικής ε, Ένωσης. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου δείχνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης στην Αφρικανική αυτή χώρα. Αλλά δεν έχουν ε, προταθεί συγκεκριμένα μέτρα για να χαιτιστεί η τραγωδία που πλησιάζει. Θα σας δώσω λοιπόν το λόγο για την ε, εισαγωγή και μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση με τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. President. Um, it's a pleasure to be E Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι ξανά στην Επιτροπή σας. Ξέρω πως ε, για πολλούς από εσάς ξεκινούν οι διακοπές. Εύχομαι λοιπόν καλά Χριστούγεννα και καλή ξεκούραση. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μία ενημέρωση για το τι έγινε στο Συμβούλιο Εξωτερικών και θα καλύψω κάποια θέματα, όχι όλα, γιατί θέλω να αφιερώσω και χρόνο στο να απαντήσω στις ερωτήσεις σας και στο να συζητήσουμε. Αλλά θα καλύψω τα βασικά. Ξεκίνησε το Συμβούλιο και κλεισμένο των θυρών και μπόρεσα έτσι να ενημερώσω τους υπουργού για το αποτέλεσμα των ε, συνομιλιών με το Ιράν. Συνομιλίες ε, στις οποίες συμμετέχω εδώ και τρία χρόνια και θα μάθατε πως 20 ε, με 24 Νοεμβρίου καταλήξαμε σε ένα κοινό σχέδιο δράσης που είναι πραγματικά ένα πρώτο βήμα για μια μακροπρόθεσμη συνολική λύση η οποία θα διασφαλίσει πως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα είναι ειρηνικό. Καλύπτει μέτρα αμοιβαίου χαρακτήρα και από το Ιράν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύν τους τρεις. Θεωρώ πως η συμφωνία της Γενέβης ήταν πραγματικά μια σημαντική διπλωματική επιτυχία. Τώρα πρέπει να περάσουμε στην εφαρμογή. Χτες συνάντησα τον πρέσβη, τον κύριο Αράτσι, υφυπουργό εξωτερικών, ο οποίος ε, συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις και θα δείτε πως οι διαπραγματεύσεις ε, επιτεχνικών ζητημάτων που είχαν σταματήσει την προηγούμενη εβδομάδα θα επαναληφθούν την Πέμπτη. Επίσης, ε, Συζητήσαμε και με τον Υπουργό, τον ε, κύριο Ζαρίφ, ε, το πώς όταν θα περάσουμε στην εφαρμογή θα ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις για μια συνολική, ελπίζω, λύση. Αντιλαμβάνεστε όλη την ευαισθησία της ε, διαδικασίας. Το μόνο που θα πω είναι πως προσωπικά εγώ και βεβαίως εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύω να ολοκληρώσω το έργο αυτό, εάν κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Επίσης είδαμε και τις πτυχές της εξωτερικής πολιτικής της ε, διεύρυνσης. Ε, Απέσλαμε μια επιστολή η οποία εξέθετε τα αποτελέσματα της διαδικασίας Σερβίας Κοσφοπεδίου και για μένα ήταν ιδιαίτερη ευχαρίστηση το ότι συμμετείχα στην διαδικασία αυτή. Ήμουν στην 20η συνάντηση, συναντήσεις οι οποίες καμιά φορά διαρκούσαν μέχρι και 14 ώρες, 14 συναπτές ώρες. Τα αποτελέσματα βεβαίω είναι φανερά σε όλους, καμιά φορά ε, υπέρευναν και τι προσδοκίε μου, π.χ. όσον αφορά τι εκλογέ στο Βόρειο Κοσμοπέδιο και εδώ πέρα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ρομπέρτο Γκαλτιέρη για την ε, εξαιρετική δουλειά που έκανε στην αποστολή παρατήρηση των εκλογών υπό ε, πολύ δύσκολε συνθήκε και τον ευχαριστώ. Την επόμενη μέρα στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων υιοθήσαμε το διαπραγματευτικό πλαίσιο για την ε, Σερβία και αποφασίσαμε να ξεκινήσουν οι δεξιακέ διαπραγματεύσει τον Ιανουάριο του 14 αναμένω και το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επικυρώσει αυτή την απόφαση. Εμείς θεωρούμε πως αυτό δεν είναι μόνο ένα σημαντικό μήνυμα για την Σερβία αλλά για ολόκληρη την περιοχή. Ελπίζω επίσης πως η Συμφωνία Σύνδεσης και Σταθεροποίησης, οι σχετικές διαπραγματεύσεις δηλαδή για το Κοσμοπέδιο θα ολοκληρωθούν το 2014. Θεωρώ πως το Κωσοπέδιο και η Σερβία είναι ένα μοντέλο το οποίο πρέπει να εμπνεύσει τα υπόλοιπα Δυτικά Βαλκάνια για να λύσουν τα ανοιχτά ζητήματα και να προχωρήσουν στο μέλλον. Και βεβαίω ε, είναι αμφισβήτη τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς ενέπνευσε τους Πρωθυπουργού ε, και τις διαπραγματευτικές ομάδες για να συμφωνήσουν. Για την Αλβανία το Συμβούλιο αποφάσισε να στείλει ένα θετικό μήνυμα να αναγνωρίσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και να υιοθετήσει κάποια συμπεράσματα τα οποία πάλι θα καταλήξουν σε ένα καθεστώς 20 χώρας ε, μέσα στο 2014, κάτι το οποίο βεβαίως θα συνεισφέρει και στην περιφερειακή σταθερότητα. Αναμενόμενο είναι πως συζητήσαμε αρκετά την Σύνοδο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στο Βίλνιους, η οποία είχε συγκεκριμένα και ουσιαστικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα όσον αφορά την μονογραφή των συμφωνιών σύνδεσης με Μολδαβία και Γεωργία. Και βεβαίω υπάρχει αυξανόμενη στήριξη για τις δύο χώρες, αλλά οπωσδήποτε μας απασχόλησαν και οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Όπως ξέρετε ήμουν στο Κίεβο την προηγούμενη εβδομάδα ε, συναντήθηκα δύο φορές με τον πρόεδρο τον κύριο δύο φορές με εκπροσώπους αντιπολίτευση, με κοινωνία των πολιτών, με τρεις πρώην προέδρους και επίσης ε, και στην ε, πλατεία την κεντρική ήμουν παρούσα. Επίσης Είπαμε πως σκοπεύουμε να υπογράψουμε την Συμφωνία Ζώνης Ελευθερίου Εμπορίου μόλις έχουν εκπληρωθεί οι συνθήκες. Βεβαίως ε, θεωρούμε πως έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για το μακροπρόθεσμο οικονομικό μέλλον της Ουκρανίας. Αλλά και βραχυπρόθεσμα θα υπάρχουν ωφέλη και πέραν όλων των άλλων θα στείλει το μήνυμα στις διεθνείς αγορές και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στην οικονομία της χώρας και βεβαίω αποτελεί και ένα υπόδειγμα μεταρρυθμίσεων. Οι Υπουργοί βεβαίως ήταν θετικοί όσον αφορά την ε, στήριξη που υπάρχει από τόσους πολλούς στην Ουκρανία για την σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως φάνηκε τις ε, τελευταίες εβδομάδες και ο κ. Γιάννου Κόβιτς ε, επανέλαβε την επιθυμία του να υπογράψει την συμφωνία και συζητήσαμε λεπτομερώς όλες τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ουκρανία. Βεβαίως, είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε για να βρεθεί ένας τρόπος να ξεπεραστεί το αδιέξοδο. Χτες έλαβα μια επιστολή από τρεις ηγέτες της αντιπολίτευσης ε, όπου εξέθεταν τις ιδέες τους και κατέστησα σαφές πως και εγώ και άλλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως έχουμε κάθε διάθεση να βοηθήσουμε στον διάλογο εάν κάτι τέτοιο ε, μπορεί να βοηθήσει βεβαίως ξεκαθάρισα πως θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα του συνέρχεστε οι πολίτες της Ουκρανίας, να μπορούν να εκφραστούν, να, μην υπάρχει βία, να ερευνηθεί η άσκηση βίας μέχρι στιγμής και βεβαίως να απελευθερωθούν οι κρατούμενοι διαδηλωτές και να επιληθεί η πολιτική αυτή κρίση για να προχωρήσει η χώρα. Μιλήσαμε για την νότια γειτονιά μας και ειδικά την Συρία, καθώς υπάρχουν δύο πτυχές που μας απασχολούν. Η πρώτη είναι η ανθρωπιστική κατάσταση, η οποία είναι τραγική. Η κυρία Γεωργίευα συναντήθηκε σήμερα με υπηρεσίες του ΟΗΕ και γνωρίζουμε πως τεράστια έκκληση του ΟΗΕ ε, είναι μόνο ένα μέρος της προσπάθειας που απαιτείται για τους ανθρώπους αυτούς που αυτή τη στιγμή υποφέρουν όχι μόνο στη Συρία αλλά και στις γειτονικές χώρες και σε κράτη-μέλη της Ένωσης όπου αναζητούν ε, καταφύγιο αυτοί οι άνθρωποι και πιθανώς και άσυλο. Η άλλη πτυχή βεβαίως μας απασχόλησε είναι η Γενεβίδη Ο Πιερβιμόν μόλις ήρθε από μια συνάντηση με τον Λαχτάρ Μπραχήμη και συζήτησαν τις προοπτικές ε, μιας, ε, ενός δεύτερου γύρου στη Γενέβη. Θέλουμε βέβαια να υπάρξει ένας ρόλος κοινωνίας των πολιτών και βεβαίω θέλουμε να εκπροσωπούνται και γυναίκες στις αντιπροσωπείες αυτές. Γνωρίζω πως ο Πιέρ το έθεσε αυτό στον Λαχτάρ Μπραχήμι, ο οποίος συμφωνεί και πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξουμε τις γυναίκες για να είναι παρούσες στη Γενέβη. Όχι στο περιθώριο, αλλά στην ουσία των συζητήσεων. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε για να συνεχιστεί η περιφερειακή συνεργασία, να στηρίξουμε τις διπλωματικές προσπάθειες, να συνεχίσουμε τις δικές μας διπλωματικές επαφές, όχι μόνο με στους ανθρώπους εντός Συρίας αλλά και εκτός και σε ολόκληρη την περιοχή όπου οπωσδήποτε ε, βρίσκεται η λύση. Επίσης, αναμένουμε να δούμε το τι θα γίνει στο μέτωπο της καταστροφής των χημικών όπλων, ε, όπου τα πράγματα πηγαίνουν καλά, αρκετά κράτη-μέλη έχουν προσφέρει ε, στήριξη στο μέτωπο της επιμελητίας. Επίσης, αναμένουμε να θα γίνει με την αποστολή την διεθνή για να ολοκληρωθεί εκεί πέρα η καταστροφή των όπλων. Θα αναφερθώ τώρα και στην κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία η οποία είναι ανησυχητική. Πρέπει να αντιδράσουμε ανησυχητικά, συνεργαζόμαστε στενά με την Γαλλία και βεβαίω είναι ευπρόσδεκτη η παρέμβασή τους. Έχουμε δώσει 50 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουμε τη δουλειά που γίνεται εκεί πέρα και βεβαίως και αρκετή ανθρωπιστική βοήθεια, άλλα 18,5 εκατομμύρια ευρώ την Δευτέρα. Αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να αντιμετωπιστεί η κρίση και να βοηθούν οι άνθρωποι της χώρας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά είναι επίσης κάτι το οποίο συζητάμε με τους Αφρικανούς εταίρους μας για να υπάρχει πιο άμεση αντίδραση σε τέτοιες κρίσεις. Αν με βεβαιώσετε ότι γίνεται την, ε, στην Αφρική, πρέπει να σα πω πως με απασχολεί και το νότιο Σουδάν αυτή τη στιγμή, στη Τζούμπα και αλλού, όπου συνεργαζόμαστε στενά με την ε, εκεί αντιπροσωπεία μας. Υπάρχει μια συνάντηση ξανά της πλατφόρμας διαχείρισης της κρίσης για να δούμε το τι μπορούμε να κάνουμε. Και τέλος κύριε Πρόεδρε, μεταξύ άλλων πραγμάτων θα ήθελα να αναφέρω την ε, ομάδα εργασίας για την Μιανμάρ Βυρμανία την οποία βεβαίως ενημερώσαμε και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την στήριξη που μας παρέχει. Είχαμε και συνάντηση στην χώρα, μια διήμερη συνάντηση με τον Πρόεδρο Τανσίν και με την κυρία Μξανσούντζη, κάτι το οποίο νομίζω είναι πολύτιμο και για το λαό της χώρας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα έχουμε τον πρώτο γύρο ερωτήσεων με τους συντονιστές. Δύο λεπτά δικαιούται ο κάθε συντονιστής. Πρώτος ο κύριος Αλαφράγκα. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε κυρία Υπατή εκπρόσωπε και αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όντως, ήσταν ε, πολύ άσχολοι το τελευταίο καιρό και σας στείλαμε συγχαρητήρια μέσω των ε, συνεργατών σας για το αποτέλεσμα των ε, διαπραγματεύσεων με το Ιράν για τα πυρηνικά και περιμένουμε και τις εξελίξεις του επόμενου εξάμεινου. Θα ήθελα να αναφερθώ στην κατάσταση στη Συρία και τι προπτικές ε, διανοίγονται για τη δεύτερη γύρο διαπραγματεύσεων στη Γενέβη που θα ξεκινήσουν 22 Ιανουαρίου. Είναι τραγικές ε, οι συνθήκες στις γειτονικές χώρες, ιδιαίτερα στο Λίβανο. Είδα και διάβασα τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών. Είναι πραγματικά μεγάλη αστάθεια. Φυσικά μας υποσχολεί και η κατάσταση στην Ουκρανία. Και η πρώτη μου ερώτηση αφορά την αξιολόγηση που θα ήθελα να κάνετε για τις ε, χθεσινές συμφωνίες της Ουκρανίας με τη Ρωσία που αφορούν κάποια χρηματοπιστωτικά θέματα, αφορούν την τιμή του φυσικού αερίου και αν πιστεύετε ότι οι συμφωνίες αυτές ε, προϋποθέτουν ε, σε μεταγενέστερο διάστημα και την σύναψη Τελωνιακής Ένωσης είδαμε και την προσωπική σας δέσμευση και με την επίσκεψη στο Κίεβο. Προσφερθήκατε και διαμεσολάβηση. Και μάλιστα αυτό περιλαμβάνεται και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρείτε ότι αυτή η πρότασή σας για διαμεσολάβηση θα ληφθεί υπόψη από τις αρμόδιες αρχές της χώρας. Και τέλος δύο ερωτήσεις. Πρώτη, πώς αξιολογείτε τα συμπεράσματα του Υπουργείου Γενικών Υποθέσεων, του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων για την αναθεώρηση των μέσο και μακροπρόθεσμη των εργασιών της ΑΕΔ. Βέβαια θα είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, αλλά με ενδιαφέρει να μάθω αν πιστεύετε κατά πόσο έχετε περιθώριο μέχρι στο ολοκληρώσει τη θητεία σας ή κάτι τέτοιο θα παραπευθεί στο διάδοχό σας. Έχετε πολύ σημαντικές αρμοδιότητες και πολλές ευθύνες, αλλά μην ξεχνάτε και τη Λατινική Αμερική. Τον Ιανουάριο που ε, μας είχατε συνοδεύσει στην διάσκεψη κορυφή του Σαντιάγου, είπαμε ότι θα κάνουμε αναθεώρηση των ε, συμφωνιών σύνδεση με το Μεξικό και τη Χιλή. Δεν έχουν προχωρήσει όμως τα πράγματα. Ελπίζω να έχουμε σχετικά σύντομο διάστημα τις διαπραγματευτικές ε, κατευθυντήρες γραμμές. Ευχαριστώ η κυρία Γκόμες εκ μέρους των Σοσιαλιστών για δύο λεπτά. Να σας συγχαρώ για την επιτυχία στο Ιράν, για το Ιράν το Ιράν ε, βεβαίως ενδιαφέρεται πολύ για την κατάσταση στη Συρία. Εμπλέκεται και στη συνάντηση με τη Γεωργίευα και τον Αντώνιο Γκουτιέρεθ και οι δύο είπαν ότι πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να καταλάβουν ότι είναι αδύνατη η στρατιωτική λύση. Ορισμένοι δεν το έχουν καταλάβει ακόμη. Όπως ε, οι Σαουδιανοί, οι Τούρκοι, οι Κατάροι. Τι τους λέει σε αυτούς τους εμπλεκόμενους η Ένωση. ούτως ώστε να έρθουν όλοι στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων Γενέβη 2 για την Ουκρανία. Θα ήθελα να ακούσω την απάντησή σας στην ερώτηση Αλανφράκα για τις οικονομικές επιπτώσεις της κατάστασης και τη συμφωνία που υπέγραψαν με την Ρωσία και ιδιαίτερα εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε τις ενέργειές σας ε, οποιασδήποτε ενέργειες πρέπει να γίνουν για την Ουκρανία που προκαλεί τόσες διαφορές απόψεων. Τέλο, για την Αφρική. Είπατε πώς έχει κατάσταση, πόσο ανησυχητική είναι στην κεντροφρικανική Δημοκρατία, όπου από τη Δύση είναι μόνη τη η Γαλλία, Νότιο Σουδάν. Θα μπορούσα να φερθώ και στο Μαλί, τη Γουινέα Μπισάου, όπου βλέπουμε ότι καταραίει το κράτος. Βλέπουμε τρομερή κατάσταση. Το πορτογαλικό αεροπλάνο αναγκάζεται να πάρει ανθρώπους ε, με ψεύτικα διαβατήρια και αυτό το κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Θα έπρεπε να έχουμε ενισχύσει αντί να μειώσουμε τις προσπαθίες μας. Πού είναι λοιπόν η εξωτερική μας πολιτική, προς τα πού πάει. Παίρνουν τις σωστές αποφάσεις οι Υπουργοί. Στο τελευταίο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων καταφέρατε να ξαναδείτε το θέμα των αποστολών της κοινή πολιτικής εξωτερικών και άμυνας, γιατί το θέμα είναι να υπάρχει μια ενοποιημένη αντιμετώπιση και πολιτική και στρατιωτική για στρατηγικές ε, ε, και κράτους δικαίου. Πού πάμε. Κάτσουν δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Εκ μέρους ε, της ομάδας ALDE θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για την ε, επιτυχία που, τις επιτυχίες που έχετε σημειώσει. Η πολιτική αυτή, η εξωτερική πολιτική της Ένωσης ε, υπάρχει και είναι αναγνωρίσιμη στην Ευρώπη και παντού στον κόσμο χάρη σε εσά. Είστε πολύ ε, σημαντικός παράγων Πολύ σημαντικότερη είναι η δράση σας από αυτή που αναμένανε πολύ όταν αναλάβατε. σε συγχαίρω και εσάς και το προσωπικό σας για το Ιράν τώρα. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που να μπορούν να εφαρμόσουν τις αποφάσεις ε, επιτόπου και να ε, εφαρμόσουν έτσι τις στρατηγικές μας αποφάσεις. Και για τα Δυτικά Βαλκάνια. Επίσης να σας συγχαρώ. Εσείς ο Ντάζιτς και ο Χάζιμ Τάτσι είστε η καλύτερη τρόικα η πιο περίφημη που θα μπορούσε να υπάρξει στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στα Δυτικά Βαλκάνια. Θα ήθελα λοιπόν να βρείτε και σε άλλες περιοχές του κόσμου δύο τέτοιους εταίρους για να έχουμε παρόμοιες δράσεις μια τρόικα στην περίπτωση για παράδειγμα της Ουκρανία. Μια τρόικα λοιπόν χρειαζόμαστε σε κάθε περιοχή που να γνωρίζει τις στρατηγικές προκλήσεις, να μπορεί να συνεργάζονται τα μέλη ανάμεσά τους και να έχει εμπιστοσύνη στη δράση της. Σας συγχαίρω λοιπόν και για το Κωσυφοπέδιο και τη Σερβία. Αλλά, να σας πω ακόμη, ότι είναι σημαντική μέρα σήμερα, γιατί το Μαυροβούνιο ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις. όχι μόνο είναι η πρώτη χώρα από την περιοχή που άνοιξε τα κεφάλαια 23 και 24, αλλά και τα κεφάλαια 5, 6 και 20. 6, 26 δηλαδή δημόσια συμβόλαια και καταπολέμηση της διαφθοράς. Είναι πολύ σημαντικές προοπτικές για να επιτευχθεί εναρμόνιση. Σας συγχαίρω επίσης για τη Μολδαβία και τη Γεωργία και για την Ουκρανία συγκεκριμένη ερώτηση. Ο κύριος Πούτιν ε, παίζει βεβαίως το ρόλο του. Είναι βεβαίως ε, ένας ρόλος στην παγκόσμια σκηνή. Γι' αυτό εμείς πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί στην αντιπαράθεση. Τι προτίθεστε να κάνετε γι' αυτό. Τελευταία ερώτηση. Συστημική διαφθορά. Είναι πρόβλημα στην Ουκρανία. Η δημοκρανία έχει απαχθεί. Θα ήθελα να μου πείτε θα κάνετε γι' αυτό. Κρόμπερκ, ε, δύο λεπτά, ε, παρακαλώ. Παρακαλώ να σέβεστε το χρόνο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ομιλητέ που έχουν ζητήσει το λόγο. Και θα κλείσω το κατάλογο. Θα ήταν αδύνατο να απαντήσει η κυρία Άστον. Ευχαριστώ. Συμφωνώ και εγώ με όσους συνεχάρισαν για το έργο σας, κυρία Βαρόνια Άστον. Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ιράν μόλις επέστρεψε από τη χώρα αυτή και έγιναν πολλές συζητήσεις εκεί με βουλευτές, με μη κυβερνητικέ οργανώσεις και με εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερικών στην Τεχεράνη. Και μάλιστα βρεθήκαμε στην Τεχεράνη τη στιγμή που βγήκαν ε, νέες ειδήσει στον παγκόσμιο τύπο ε, και οι αντιδράσεις ε, του Ιράν για τα σχόλια που έγιναν στις ΗΠΑ ήταν πολύ αρνητικά και φυσικά κατηγόρησαν τους Αμερικανούς. Και μάλιστα υπήρχε μια ένταση μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργού Εξωτερικών και των βουλευτών στο Ιράν, γιατί ο Υπουργός Εξωτερικών μας έδωσε την εντύπωση ότι αυτοί οι κατάλογοι του Υπουργείου Οικονομικών ε, δεν παραβίαζαν την Συμφωνία της Γενέβης, ε, τουλάχιστον ως προς το πνεύμα της και ότι θα συνεχιστούν οι σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ενώ οι βουλευτές του Ιράν ήταν επικριτικοί. Θεώρησαν αυτή τη δημοσίευση των καταλόγων ως παραβίαση της συμφωνίας και κατηγόρησαν τις Ηνωμένε Πολιτείε και άσκησαν ε, επικρίσεις στον Υπουργό Εξωτερικών. Υπήρχε μία ένταση. Δεν έγινε συζήτηση για το κατά πόσο οι παλιές ή οι νέες ε, ισχύουν ή δεν έγινε συζήτηση για τις, για λεπτομέρειες. Ο Υπουργός Εξωτερικών λοιπόν ακολουθούσε αυτή τη γραμμή ενώ οι βουλευτές ε, που ήταν πιο σκληροπυρηνικοί ήταν πιο επικριτικοί. Ποια είναι η δική σας γνώμη, η κατάλογοι του Υπουργείου ε, Οικονομικών των ΗΠΑ πώς Πώ αντιμετωπίστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι εντύπωση προκάλεσαν και πώ θα του χαρακτηρίζατε. Ο κύριο Στάνοκ. Ευχαριστώ, Λέδη Άστον. Σας συγχαίρω. Πολύ καλή χρονιά για εσά. Οι συμφωνίε Βελιγράδιου και Πριστίνας και οι συμφωνίε για τη Γενέβη και οι συμφωνίε για τι πυρηνικέ φιλοδοξίε του Ιράν όσον αφορά τον εμπλουτισμό του ουρανίου. Ουκρανία τώρα. Είπατε ότι ο κύριο Γιανουκόβιτ, σας είπε εσάς ότι θέλει να υπογράψει τη Συμφωνία Σύνδεσης. Μα δεν συμβιβάζεται με αυτά που λέει στις επιπτώσεις, με τις επισκέψεις του στο, στη Μόσχα και στο Σότσο, όπου ε, ε, ε, έκαμψε τη μέση στην Ρωσία και είπε ότι θέλει να υπογράψει συμπορικές συμφωνίες μαζί τους. Αλλά εν πάση να επανέλθω σε αυτό που είπε η Άννα Γκόμες. Τι νέα καρότα θα μπορούσαμε να έχουμε για να ε, τους βοηθήσουμε να στραφούν προς εμάς. Και τι θα γίνει αν ε, υπάρξει βία για να φύγουν οι άνθρωποι από το Μαϊντάν. Θα μπορούσε τότε να έχουμε επιπτώσεις, ε, κυρώσεις όπως αυτές που επιβάλαμε στη Λευκορωσία. Και βεβαίως η Ρωσία προσπαθεί αποφασισμένα να επανέλθουν οι πρώην οι πρώην Σοβιετικές χώρες ε, στη σφαίρα επιρροής της. Θα εξακολουθήσουμε να έχουμε σχέσεις τέτοιες με τη Ρωσία εάν υποστηρίξει η Ρωσία τις προσπάθειες ε, Γιαννουκόβιτς να ξεκαθαρίσει την κατάσταση των Μαϊντάν δια της βίας για το Ιράν. Είναι σαφές ότι το Ιράν ε, ήταν αρκετά δύσκολος πελάτης στο παρελθόν. Ξεγλιστρούσε. Αν σε μερικού μήνε διαπιστώσουμε ότι έχουν παραβιάσει το περιεχόμενο τη συμφωνία, Πώς θα ε, επανεπιβάλλουμε τις ε, κυρώσεις, τι θα κάνουμε. Τώρα που έχουμε ξεπαγώσει όλες τις πιστώσεις, άρα θα επιστρέψουν στο Ιράν και για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα έπρεπε να κινητοποιηθούν οι ομάδες μάχης της εξωτερικής μας άμυνας και ασφάλειας. Ποτέ δεν έχουν ε, αξιοποιηθεί, δεν θα μπορούσαν να βοηθήσουν να σταθεροποιηθεί αυτή η χώρα. Ευχαριστώ. Έχω και εγώ μια ερώτηση, Λέει Άσταν για τη Συρία. Σε πολλές περιοχές της χώρας ε, φαίνεται ότι ενισχύονται οι Ισλαμικές εξτρεμιστικές δυνάμεις και η Αλκάιδα επιβάλλει το δικό της νόμο. Ξεκινώντας από τα στοιχεία αυτά, κάποιοι παρατηρητές ε, ζητούν να συνεχίσουμε τις συζητήσεις ε, με, τη, με το καθεστώς του Ασάτ και ο Ράιν Κρούγκερ πρέσβης στο Ιράκ, ε, Αμερικανός, είπε σε ένα άρθρο στους New York Times ότι ίσως θα ήταν καλύτερα να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, οι συνομιλίες με το καθεστώς του Ασάτ και ότι καλύτερα ο Ασάτ παρά οι τζιχαντιστικές εξτρεμιστικές ομάδες που θα μπορούσαν να επικρατήσουν στη χώρα τι συνιστά η εξέλιξη αυτή, πολιτική αποτυχία ή επίδειξη πολιτικού ρεαλισμού. Ποια είναι η γνώμη σας και η αξιολόγησή σας. Ευχαριστώ. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις. Να ξεκινήσω με τις ερωτήσεις του κυρίου Σαλαφράγκα και να σας ευχαριστήσω όλους θερμά για τα ευγενικά σας λόγια ε, για την Σερβία, το Κωσυφοπαίδιο και το Ιράν. Προσδοκίες τώρα για τη Γενέβη 2. Εγώ πιστεύω ότι βρισκόμαστε στην αφετηρία της διαδικασίας. Δεν έχω καμία προσδοκία ότι θα διεκπαιρεώσουμε τις διαδικασίες αυτές σε μία μόνο μέρα στη Γενέβη. Θα ξεκινήσει ο διάλογος που θα οδηγήσει καταρχήν σε μία κεχηρία, προκειμένου να φτάσει στη χώρα η ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό τώρα. Να σταματήσει ο πόλεμος και να φτάσουν τα τρόφιμα το νερό και μια φροντίδα στον άμαχο πληθυσμό. Και ελπίζω ότι με τις προσπάθειες που κάνει ο κύριος Μπραχήμη και τα διαβήματα προς όλες τις κατευθύνσεις θα καταφέρουμε να φέρουμε στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων όσους ασκούν κάποια επιρροή ε, για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Θα είναι βέβαια μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Είναι προφανές από ό,τι βλέπουμε, διαβάζουμε και από τις επαφές που είχαμε γιατί έρχονται πολλοί και διάφορες Βρυξέλλες και έχουμε επαφές σε όλο τον κόσμο για το θέμα αυτό, αλλά θα πρέπει επιτέλους ε, να δοθεί το αναρκτήριο λάκρισμα. Αν δεν υπάρξει η αρχή, δεν θα έχουμε καμία ελπίδα να καταλήξουμε κάπου. Και όντως είναι πολύ έθραυστη κατάσταση στο Λίβανο και από πολιτική άποψη, αλλά με 25% του πληθυσμού να είναι σήμερα πρόσφυγες από τη Συρία, η διαχείριση της κατάστασης είναι εξαιρετικά δύσκολη για το Λίβανο. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες αλλά και την πολιτική διαδικασία προκειμένου να ε, μπει στα σκαριά και η νέα κυβέρνηση. Τώρα για την Ουκρανία. Πολλές ερωτήσεις ε, για το θέμα αυτό και από τον κύριο Τάνοκ. Επαναλαμβάνω αυτά που μου είπε ο κύριος Γιαννουκόβιτς, επανειλημμένος δήλωσε επανειλημμένω ότι θέλει να υπογράψει τη συμφωνία αυτή και ότι όλη η πολιτική του σταδιοδρομία στηρίχθηκε στην υπογραφή αυτή τη συμφωνία. Και είπε ότι αυτή είναι η επιθυμία του και η πρόθεσή του. Τώρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτά που έλαβε. Αν τα εννοούσε είναι άλλο θέμα. Πάντως αυτό δήλωσε επίμονα και επανειλημμένος. Τώρα υπάρχουν όμως κάποια βραχυπρόθεσμα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και Εμεί δεν διαφωνούμε ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια καλή σχέση με τη Ρωσία. Δεν αποκλείται το ένα το άλλο. Είναι συμπληρωματικέ οι σχέσει ε, και με τη Ρωσία και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εμεί θέλουμε καλέ ε, συμφωνίε με την Ρωσία. Έχουμε εμπορική συμφωνία. Αυτές, οι καλέ σχέσει θα συνεχιστούν. Γιατί υπάρχουν παρεξηγήσει και παραπλάνηση, παραπλανητική ενημέρωση για τις, συμφων... για τις συνέπειες της συμφωνίας για μας. Θα πρέπει να ενημερώσουμε καλύτερα για τις συνέπειες. Αν δούμε την οικονομική ανάπτυξη που αναμένεται στην Ουκρανία ε, μακροπρόθεσμα, ε, το θετικό αποτέλεσμα και ο αντίκτυπος θα φτάσει και στη Ρωσία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ε, θα έχουμε κατά ανάγκη αρνητικό αποτέλεσμα. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν με τρόπο που θα υποστηριχθούν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την στήριξη αυτή και δραστηριοποιούνται στην Ουκρανία και ήδη υπάρχουν προσφορές προς την Ουκρανία από πολλές και διάφορες πηγές. Από φορείς που είναι έτοιμοι να επενδύσουν στο μέλλον της Ουκρανίας. Οπότε τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα που όντως υπάρχουν μπορούν να επιληθούν και μάλιστα στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας. Επίσης, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι δεν άκουσα τίποτα και το είπα και σε συνέντευξη τύπου στην Ουκρανία. Τίποτα από αυτά που άκουσα δεν ε, μου δημιούργησαν υπόνοιες ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην ουσία των προσπαθειών μας και ότι θα εμποδιστούμε στην διεκπαιρέωση αυτών των προσπαθειών. Σε ό,τι αφορά την ε, παρεξέταση και αναθεώρηση της ΕΙΕΔ, υπάρχει το βράχι, μέσο και μακροπρόθεσμο θέμα και μια διαφοροποίηση. Εμείς θέλουμε πρώτα να επιλύσουμε τα βραχυπρόθεσμα ζητήματα και να τα διεκπαιρεώσω στη διάρκεια της δικής μου θητείας. Γιατί για τα μακροπρόθεσμα θα χρειαστούν και κάποιες νομοθετικές αλλαγές, γιατί βρισκόμαστε ουσιαστικά στα σπάργανα της ε, υπηρεσίας αυτής. Και φυσικά θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή το συντομότερο δυνατόν. Και σίγουρα θα γίνουν συζητήσει με κράτη-μέλη που έχουν και διεστάμενε απόψει. Το Συμβούλιο θα πρέπει να λάβει τι αποφάσεις του με βάση την κρατούσα γνώμη, τη συνένεση που υπάρχει. Και εκεί ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγης τα πράγματα και θα βοηθήσει και το διάδοχό μου να λάβει υπόψη και τις δικές του ανησυχίες. Γιατί όσο περνάει ο χρόνος θα αναπτύσσεται η ΕΕΔ και θα ανακύψουν και άλλα θέματα. Αυτά ως προς την αναθεώρηση. Ευελπιστώ ότι δεν θα μπει ε, στα συρτάρια το έγγραφο της αναθεώρησης, αλλά θα προκαλέσει ενδιαφέρον και ελπίζω ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι πραγματικά με αυτή την ανάμειξη θα κάνουμε και κάτι διαφορετικό. Ο πρόεδρος Μπαρόσο μόλις επέστρεψε από την Κολομβία και το Παναμά. Δεν ξεχνούμε τη Λατινική Αμερική σε καμία περίπτωση. Θα συνεχίσουμε να ε, αναπτύσσουμε τις σχέσεις μας και ελπίζω στις αρχές του επόμενου έτους να διαμορφώσουμε, να οριστικοποιήσουμε και κάποιες ιδέες που έχουμε για το Μερκοσούρ. Και σημαντικό θα ήταν να έχουμε εξελίξεις. Πάντως, ένας από τους λόγους που πήγε ο κύριος Μπαρόζο εκεί είναι ακριβώς για να δείξει την υποστήριξή μας προς τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στη Λατινική Αμερική και ευελπιστούμε ότι θα συνεχιστούν. Και θα δούμε αν θα στείλουμε και εκπρόσωπο στην α, ε, α, ε, ανάληψη των καθηκόντων της α, ε, νέας πρόεδρου της Χιλής κυρίας Μπασιλέ. Είναι δύσκολα πάντως τα πράγματα όταν επικεντρωνόμαστε σε συγκεκριμένα θέματα γιατί το Ιράν, το Κωσυφοπαίδιο ήταν πολύ σημαντικά ζητήματα που απέσπασαν την προσοχή μας για πολύ καιρό αλλά δεν ξεχνούμε και τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες περιοχές. Άννα Γκόμες, Συρία. Τι λέμε στους συνομιλητές μας. Το θέμα είναι ότι την ειρήνη δεν την συμφωνούμε με τους φίλους, αλλά με τους εχθρούς. Είναι σημαντικό λοιπόν οι συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις να μπορέσουν να λάβουν κάποιες αποφάσεις. Και με πολλούς και διάφορους τρόπους προσπαθούμε να αναμίξουμε χώρες και ομάδες ε, που δεν βρίσκονται κατά ανάγκη στον πυρήνα των διαπραγματεύσεων. Στη Γενέβη έχουμε έναν πυρήνα συμμετεχόντων και έχουμε και άλλες ε, ομάδες και χώρες που συμμετέχουν. Ο κύριος Μπραχήμη είναι ιδιαίτερα προσιλωμένος στο θέμα αυτό και καλό θα ήταν να τον υποστηρίξουμε για να βρει τους σωστούς συνομιλητές και να τους φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Για την Ουκρανία τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό που έχει κάνει ήδη, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε το παρόν στην Ουκρανία, έστειλε μήνυμα στους βουλευτές, στην κυβέρνηση. Αυτό θα πρέπει να συνεχίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει, να στέλνει αυτά τα μηνύματα και είναι σημαντικό να έχετε τακτικές επισκέψεις στην Ουκρανία. Για τη Γουενέα Μπισάο θα πρέπει να αποκατασταθεί το κράτος δικαίου στη Γουενέα Μπισάο, κάτι που είναι δύσκολο. Και υπάρχει και το θέμα της Πορτογαλικής Αεροπορικής Εταιρείας. Το συζητήσαμε με τον Πορτογάλο Υπουργό στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, ε, Εξωτερικών Υποθέσεων. Περιμένουμε τη νέα κυβέρνηση και ελπίζω οι ένοπλες δυνάμεις να συμφωνήσουν να εξέλθουν από την πολιτική σκηνή. Και έπα, θα το σχολιάσω αργότερα πιο λεπτομεριακά. Έχω συντάξει ένα μακροσκελές έγγραφο προκειμένου ε, να επικεντρώσω την προσοχή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στα επόμενα βήματα της ε, ΚΕΠΑ και το ποια θα είναι η παρουσία μας στην παγκόσμια σκηνή. Έχουμε καλές αποστολές, μερικές φορές αποχωρούμε από αυτές, γιατί οι αποστολές θα πρέπει να έχουν ε, μια πεπερασμένη διάρκεια. Είναι σημαντικό λοιπόν το Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό να συζητήσει και αυτά τα θέματα. Είναι ένα ζήτημα που δεν έχει ζητηθεί από το 2008. Ε, κύριε Κάτσιν, πολύ ευγενικό ο χαρακτηρισμός σας ότι ήμουν η καλύτερη τρόικα με τους εκπροσώπους της Σερβίας και του Κωσυφοπεδίου. Ελπίζω αυτά που έγιναν και οι συμφωνίες ε, εκεί να χρησιμοποιηθούν ε, και να μεταδοθούν, να γίνουν υπόδειγμα και να μεταδοθούν σε, σε όλη την περιοχή. Γιατί πραγματικά επιλύθηκαν μερικά δύσκολα πρακτικά θέματα, χωρίς ε, να καταπατηθούν οι κόκκινες γραμμές ε, των μεν των δε. Υπάρχει και το θέμα πάλι του ρόλου της Ρωσίας ε, στο ζήτημα της Ουκρανίας. Η Ουκρανία χρειάζεται ισχυρή σχέση, στενή σχέση με τη Ρωσία. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Και όταν ήρθε ο Υπουργός Λαυρόφ στο γεύμα, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, το δηλώσαμε. Ε, τα κράτη κάνουν επιλογές ε, και θα πρέπει να τις εφαρμόζουν και να δούμε τι εμποδίζει μερικές χώρες να εφαρμόσουν τις επιλογές τους ή να τις υποστηρίξουμε σε κάποια πρακτικά ζητήματα. Οι συζητήσεις που έγιναν στη Μόσχα και μου τα εξήγησε ο κύριος Γιαννουκόβιτς, ουσιαστικά στόχο είχαν τη σταθεροποίηση των τιμών του φυσικού αερίου και μία μείωση των τιμών και προσαρμογή στον όγκο του φυσικού αερίου. Και επίσης αγορά ομολόγων ε, ύψους 50 δισεκατομμυρίων από τη Ρωσία, εθνικών ομολόγων ε, της ε, Ουκρανίας. Σε, σε αμερικανικά δολάρια μιλάω όλα αυτά, αυτή η συμφωνία, δεν εμποδίζουν τη δική μας πορεία για τη σύναψη συμφωνίας με την Ουκρανία. Είπα ότι είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε τη συμφωνία. Η προεργασία έχει γίνει, εμείς είμαστε πανέτοιμοι και ελπίζω ότι και η Ουκρανία θα συνεχίσει αυτή την πορεία που ο κύριος Γιάννουκόβης, ο πρόεδρος Γιάννουκόβης, με διαβεβαίωσε ότι θα ακολουθήσει. Και αυτά τα μηνύματα επανειλημμένως έκανε θα γίνει τι επόμενε μέρε. <coughs> Κυρία Κρόνμπεργκ, μα μιλήσατε για την επίσκεψή σα στο Ιράν. Πολύ ενδιαφέρον να ακούω τι εντυπώσει που αποκομίσατε από την Τεχεράνη. Αυτή η κατάλογη του Υπουργείου Οικονομικών ε, των Ηνωμένων Πολιτειών ε, αφορούν τις προηγούμενες κυρώσεις, δεν είναι κάτι καινούριο. Το θέμα είναι ότι καμιά φορά στα μέσα εμφανίζονται, ξέρετε, νομίζω ότι οι Ιρανοί γνωρίζουν. Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις και όταν ο Υφυπουργό Εξωτερικών ε, και εγώ το συζητήσαμε, μου είπαν ότι ε, υπάρχουν καλά νέα. Οι τεχνικές ε, συζητήσεις ξεκινάνε την Πέμπτη στο, στη Βιέννη. Ελπίζω να καταλήξουν να γίνει πολλή δουλειά, ούτως ώστε η πολιτική συμφωνία να καταλήξει σε ένα τεχνικό πλαίσιο. Και γίνονται στην Βιέννη, γιατί θα συμμετάσχει ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας. Ο Χέλμουντ ήταν εκεί. Εγώ είμαι σε επαφή με τον Γενικό Διευθυντή και ελπίζω να γίνει. Κύριε Τάνοκ, είπατε ότι πρέπει να τους δώσουμε κάποια κίνητρα, κάποια καρότα. Ναι. Τώρα δεν θα αρχίσουμε τώρα πλειοδοσία με τη Ρωσία ή με κανέναν άλλον. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Κριστίν Λαγκάρτ έχουν κάνει δηλώσει, έχουν καταστήσει σαφέ ποια είναι η θέση του. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επίση θέλει να βοηθήσει την Ουκρανία. Υπάρχουν πολλέ δυνατότητε για επενδύσεις, για ανάπτυξη στην Ουκρανία, για να προχωρήσει η οικονομία. Αλλά κατέθεσα σαφές και στον πρόεδρο. Δεν είναι να πάρτε μερικά φράγκα για να δεχτείτε αυτά που λέμε. Υπάρχουν συγκεκριμένε ανησυχίε, συγκεκριμένα θέματα που είναι απόλυτα λογικό να έχει κάθε χώρα για το πώ θα αναπτυχθεί η οικονομία, πώ θα περάσει από μια κατάσταση σε άλλη. Εντάξει, είναι τομεί που μπορούμε να συζητήσουμε. Πώς θα στηρίξουμε τη βιομηχανία. Τι θα κάνουμε για τους πιο ενδεείς που μπορεί να κινδυνεύσουν γιατί δεν υπάρχει πια δίχτυα ασφαλείας. Αλλά αν δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν σε δύο τομείς που συζήτησα. Πρώτος, δυνατότητες της γεωργίας. Δεύτερον, στον τομέα της ενέργειας. Και βεβαίως υπάρχει και δουλειά που κάνουν για τις τεχνολογίες και τις υποδομές. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες για ουσιώδη ανάπτυξη της Ουκρανικής οικονομίας μέχρι ψηλωτά του επίπεδου. Αυτό σημαίνει ότι θα δώσει και στις αγορές ε, κίνητρα. Και άρα πιο πιθανό είναι ότι θα μπορέσουν να λάβουν τι επενδύσει που επιθυμούν. Αυτό είναι το μήνυμα που τους δίνω και θα συνεχίσω να το δίνω. Μου είπατε τι θα γίνει αν παραβιάσει το Ιράν τι κυρώσει. Μα εμεί ελπίζουμε να μην γίνει. Αυτή είναι η φιλοδοξία μα. Θα υπάρξει συμφωνία εφαρμογή. Πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσει και θα προχωρήσει η κατάσταση. Και από τις συζητήσεις μου με το Ιράν αυτό ακριβώς είναι το μονοπάτι που πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή βαδίζουμε και αυτός είναι ο στόχος μας. Να υπάρξει αυτό το σχέδιο εφαρμογής και κατόπιν να συνεχίσουμε την εργασία μας και να καταλήξει η εργασία μας. Μου είπατε επίσης τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για τις ε, ομάδες μάχης αρκετά δεν θεωρούσαν ότι ήταν σκόπιμο να εμπλακούν οι στρατιωτικές μας δυνατότητες αυτή τη στιγμή στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Όπως ξέρετε, προσπαθούμε να υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των 28 πριν πάρουμε τις αποφάσεις. Έτσι είναι η κατάσταση. Κύριε Πρόεδρε, εσείς με ρωτήσατε για τη Συρία. Συγκεκριμένα, για να δω, για να δω, πού το είχα. Α, ναι, ε, αν μπορούμε να συνομιλήσουμε με τον Άσαντ. Κοιτάξτε, πέρα από οτιδήποτε άλλο, ο Άσαντ και το καθεστώς του είναι ένοχοι διότι ε, σκότωσαν και δεν προστάτευσαν τεράστιο αριθμό ατόμων, πολιτών τους. Η απλή άποψή μου είναι ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο πρέπει να φεύγεις από την εξουσία. Ό,τι και αν συμβεί στο μέλλον όπως και αν ε, διαμορφωθούν και προωθηθούν και ελπίζουμε να προχωρήσουν οι συζητήσεις στη Γενέβη, πρέπει να δώσουμε στο λαό της Συρίας μια νέα δυνατότητα να έχει μια κυβέρνηση που θα φέρει ειρήνη και ευημερία στη χώρα. Αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος μας. Αυτή πρέπει να είναι η κοινή μας προσέγγιση προς τις συνομιλίες. 75% της χώρας είναι ερήπια. Τα παιδιά έχουν υποστεί τρομερά τραύματα. Υπάρχουν παιδιά λίγων ετών που έχουν ζήσει μόνο αυτή την κατάσταση. Δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν τρόφιμα, δεν υπάρχουν φάρμακα. Είναι άθλια κατάσταση και είναι τόσο κοντά μας. Και ό,τι και αν συμβεί στο μέλλον θα πρέπει οπωσδήποτε να μπορέσουν μέσα από τις τάχτες να προκύψει μια κυβέρνηση που να στηρίζεται από το λαό, που να μπορεί να βοηθήσει το λαό και όχι αυτήν την αιματοχυσία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, 12 συναδέλφους έχω εδώ που θέλω να μιλήσω, ένα μισή λεπτό για τον καθένα. Η κυρία Γκαμπριέλ πρώτη. Ευχαριστώ. Κυρία Υπάτη εκπρόσωπε, καταρχήν σας ευχαριστούμε για το έργο σας και τη συνεχή σας δέσμευση και προσήλωση και Συγχαρητήρια και για τις ε, ικανότητες ε, τις διαπραγματευτικές που δείξατε από την αρχή της ανάληψης ε, των καθηκόντων σας. Ήμουν στην Δημοκρατία του Κονγκό στην εκλογή παρατήρηση εκλογών το 2011 για τις βουλευτικές και τις προεδρικές εκλογές. Ελπίζω να συνεχιστεί η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας. Οι πρόσφατες εξελίξεις στο Κονγκό φαίνεται ότι είναι πολύ θετικές. Ε, και για την Καμπάλα ε, έχουμε τις ε, επιθέσεις κατά του RDLR. Και μάλιστα πρόσφατα είχα μια συνάντηση με τον Μαρτίν Κομπλέρ, τον επικεφαλής της Μονούσκο, μια διάσκεψη μετά από τις εκλογές, δύο χρόνια μετά από τις εκλογές, γιατί ήταν πολύ σημαντική παρουσία και φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώσαμε όμως ότι σήμερα δημιουργείται ένα παράθυρο ευκαιρίας για το Κονγκό για να σταματήσει ο κύκλος της, των, και να επανέλθει στη δημοκρατία και στη σταθερότητα. Βέβαια, φαίνεται ότι έχουμε αντιφατικά μηνύματα. Έχουμε τα Ηνωμένα Έθνη, τις Ηνωμένε Πολιτείε, τις Σκανδιναβικές χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο που ενισχύουν την παρουσία της και κινητοποιούν τους σπόρους τους στο Κονγκό. Τι κάνουμε όμως εμείς, πώς θα εξασφαλίσουμε το ρόλο του Συμβουλίου και την εμπειρογνωμοσύνη του ΕΣΕΚ ε, στην Κινσάσα για να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις στο τομέα της ασφάλειας και πώς ε, θα διασφαλίσουμε την προστιθέμενη αξία του γραφείου της ΕΣΕΚ στην κόμμα, πώς θα αξιοποιήσουμε ε, τις μέχρι, τα μέχρι στιγμής επιτέγματα μας μετά τις αποστολές και του ΣΕΚΠΟΛ. Διακοπή το μικροφόνο. 1,5 λεπτό κύριος Γαλτιέρο. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ για τις επιτυχίες σας σε πολλά θέματα, κυρίως στον διάλογο Σερβίας Κοσμοπεδίου. Ως επικεφαλής παρατηρητής είχα την δυνατότητα να διαπιστώσω πώς έχουν τα πράγματα και πόσο μεγάλες δυνατότητες έχει μια συνολική προσέγγιση όταν υπάρχει ισχυρή ηγεσία και σαφή στρατηγική. Και έρχομαι εδώ πέρα έτσι, στην εξέταση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Εμείς ε, καλωσορίζουμε την έκθεση του Ιουλίου 2013 που καλύπτει τα περισσότερα ζητήματα που αναφέρει η σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αναμένουμε τώρα και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Ήδη το είπε ο κύριος Σαλφράκη. Εγώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Πρώτον, πώς ενώ το Συμβούλιο διαχωρίζει τις ε, βραχυπρόθεσμες από τις μακροπρόθεσμες ε, συστάσεις, εμείς προσπαθούμε να δούμε πώς θα υπάρχει μια συνέχεια στην διαδικασία. όχι μόνο το τι θα κάνει η επόμενη εκπρόσωπος, αλλά και τι γίνεται τώρα. Το επόμενο σημείο στο οποίο έχουμε κάποιες διαφορές είναι πώς θα ενισχυθούν οι δυνατότητες της υπηρεσίας. Βλέπετε πώς ε, υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν μέσω μιας ε, ε, διαδικασίας η οποία εμείς θεωρούμε πως θα πρέπει να εμπλέκει περισσότερο αυτούς οι οποίοι έχουν μια πείρα και αντίληψη των ζητημάτων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Καλησπέρα σας. Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων δικαίως εκφράζει την ανησυχία του για την κρίση στην κέντροαφρικανική Δημοκρατία. Η παράγραφος 7 των συμπερασμάτων φαίνεται να υπονοεί πως ε, είναι πιθανή μια αποστολή ΚΕΠΑ αλλά οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να λάβουν τις αποφάσεις για την ε, ανάπτυξη μιας ε, μονάδας μάχης είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ελπίζω να είστε σε θέση με τον πρόεδρο Μπαρόζο να προωθήσετε μια τέτοια ε, απόφαση. Γιατί, εάν δεν είναι αποφασιστική στο θέμα αυτό. Δεν θα απογοητεύσουμε μόνο τους ανθρώπους της χώρας, αλλά θα έχουμε πλέον ερωτήματα για τον σκοπό των μονάδων μάχης. Είναι απλά διπλωματικές πυρουέτες ή υπάρχουν για να σώζουν ζωές. σας στήριξε μέχρι και ένας Βρετανός συντηρητικός και ένας φιλελεύθερος. Οι τρεις μας ίσως νομίζω κάτι θα μπορούσαμε να επηρεάσουμε στην ε, Βρετανική κυβέρνηση η οποία αποφάσισε να προβάλλει βέτο στην ανάπτυξη τέτοιων μονάδων. Σας ευχαριστώ κύριο Σούλτς για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ και εγώ την ε, Λέδη Άστον. Ευχαριστώ για την πολιτική σας δέσμευση, την καλή εργασία που κάνατε για να υπάρξει συντονισμένη ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Ο πρόεδρος Γιαννούκοβιτς πήρε την βραχυπρόθεσμη βοήθεια που χρειάζεται η χυμαζόμενη χώρα του, 50 δις δολάρια πιστώσεις από τη Ρωσία και ένα τρίτο μείωση της τιμής του αερίου. Αυτή η ρωσική υποστήριξη, μήπως ε, συνδέεται με αίτημα να κλείσουν την πόρτα στην ε, Ένωση και έγινε σαφής η διάθεση διαλόγου της Ένωσης. Δεν πρέπει να τους πούμε όμως επίσης ότι θέλουμε να παίξουμε και το ρόλο διαπραγματευτεί. Α, συγγνώμη, ότι ώστε ο γύρος διαπραγματευτών στην ε, Ουκρανία να έχει αξιοσέβαστους και σωστούς συνομιλητές. Ο κύριος Στυλ. Λοιπόν, και εγώ να συγχαρώ για τη συμφωνία για το Ιράν, το Βελιγράδι και την Πρίστινα. Αλλά είναι πρόκληση η Ουκρανία. Η Ρωσία ασκεί όλο και περισσότερη επιρροή. Όχι μόνο εκεί αλλά και αλλού. Στην Ήπειρό μας. Τα ε, πιο εκτεταμένα σύνορα της Ένωσης, είτε το πιστεύετε είτε όχι, είναι με την Βοσνία-Ερζεγοβίνη και μου φαίνεται ότι κάποιοι άλλοι που δεν είναι στην Ένωση, ε, όπως η Ρωσία και η Τουρκία, έχουν περισσότερη επιρροή στη χώρα αυτή. Δεν υπάρχει λογική πολιτική έναντι αυτού του τόσο σημαντικού τμήματος των Βαλκανίων από το οποίο τμήμα εξαρτάται η σταθερότητα των Βαλκανίων. Μπορούμε λοιπόν επιτέλους να ανασκουμποθούμε. Ξέρω ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι πρόβλημα για ορισμένα κράτη-μέλη. Δεν είναι πρόβλημα το ότι η Τουρκία έχει τόση επιρροή, αλλά για άλλου ίσω να είναι. Μπορούμε να έχουμε λοιπόν μια ε, λογική και συντεταγμένη πολιτική για τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντοκεζέρ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Άστον, σας έγραψα για να συγχαρώ για το Ιράν. Δεν θα τα ξαναπώ λοιπόν. Δύο ερωτήσεις. Συρία και Νότιο Σουδάν. Συρία. Για τη Γενέβη 2. Τι συγκεκριμένο ρόλο μπορεί να παίξει η Ένωση. Ούτως ώστε να έχουμε τη συγκεκριμένη ορατότητα όπως αυτή που είχαμε μέσω ε, της δικής σας δραστηριότητας διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Ξέρουμε ότι η δράση σας έχει συνέχεια αλλά το γεγονό, γεγονός αυτό θα τραβήξει πολύ την προσοχή των μέσων για τον Νότιο Σουδάν. Ήμουν εισηγήτρια, ψηφίσαμε μια έκθεση πρόσφατα στο Στρασβούργο, στην τελευταία Ολομέλεια, όπου τονίζουμε πόσο εύθραυστη είναι η κατάσταση και πόσο μπορεί να εκτραπεί το καθεστώς και η κυβέρνηση της Τζούμπα. Ποια είναι η ανάλυση σας, τι ακριβώς γίνεται εκεί κάτω. Τι πληροφορίες έχετε από την αντιπροσωπεία σας. Πρόκειται για πραξικόπημα. Είναι ψεύτο πραξικόπημα. Είναι κάποια νέα απαράδεκτη ενέργεια του Σαλβακύρ. Βεβαίως, ε, ίσως τον προωθήσαμε λιγάκι γιατί ήταν ο κύριος συνομιλητής μας τότε. Γι' αυτό σας ρωτάω λοιπόν τώρα. Κάναμε τόση προσπάθεια ως Ευρωπαϊκή Ένωση για να σταθεροποιήσουμε αυτή τη χώρα. Δαπανίσαμε πολλές πιστώσεις, κάνατε τεράστιες προσπάθειες, αλλά παρόλα αυτά τα αποτελέσματα δεν επαρκούν. Ήθελα λοιπόν τη γνώμη σας. Ο κύριος Βάγγελ. Ευχαριστώ. Κυρία Άστον, μετά την συνάντησή με τον πρόεδρο Γιανοκόβιτς κάνατε μια σύντομη δήλωση που συνέβαλε σε μια πιο ρεαλιστική αποτίμηση της κατάστασης στην Ουκρανία. Το τελευταίο διήμερο ακούσαμε δηλώσεις για νέο σιδηρό παραπέτασμα στην Ευρώπη, νέα φάση ψυχρού πολέμου και το καθεξής. Δεν νομίζω ότι τέτοιοι χαρακτηρισμοί θα μας βοηθήσουν να κάνουμε μια σοβαρή εμπεριστατωμένη και υπεύθυνη κρίση για την πορεία της Ουκρανίας. Πιστεύω ότι η πορεία της Ουκρανίας θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή. Είναι ευρωπαϊκή χώρα, έχει ευρωπαϊκές παραδόσεις. Αλλά δεν ευσταθεί ότι έχουμε δύο μισά στην Ουκρανία. Το ένα μισό είναι ρωσικό και το άλλο ε, ευρωπαϊκό. Έχουμε δύο μέρη, αλλά το ένα μέρος χρησιμοποιεί την Ουκρανική γλώσσα και το ανατολικό τμήμα μιλάει ρωσικά. Αλλά μόνο αυτή η διαφορά ισχύει διάβασα για κάποιες δημοσκοπήσεις που λένε ότι έχουμε περίπου ίσο αριθμό και στα δύο ε, ε, ε, ίδιο αριθμό Ουκρανών που πιστεύει στην ανατολική προοπτική και στη δυτική προοπτική της Ουκρανίας. Πάντως σας συγχαίρω θερμά για τη σύνεση που δείξατε, τη σοφία και το αίσθημα ρεαλισμού στις ε, εκτιμήσεις που κάνατε για την κατάσταση στην Ουκρανία. Ο κύριος Μιγιάν Μόν. Ευχαριστώ. Λακωνικά. Ζητώ συγγνώμη γιατί έφτασα καθυστερημένα. Δεν ξέρω αν είπατε, κυρία Άστον, για, την... για το γεύμα με τον Υπουργό Εξωτερικών Λαυρόφ. Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια τη συνάντηση με τον ε, Υπουργό Λαυρόφ γιατί έλαβε χώρα μετά τη διάσκεψη κορυφής του Βίλνιους και λίγο πριν τη διάσκεψη κορυφής με τη Ρωσία. Πώς αξιολογείτε την πρωτοβουλία της πλειοψηφίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε στο πλαίσιο της ε, έρευνας που γίνεται στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για την περίπτωση Σνόουντεν και τη μαζική παρακολούθηση από την ε, Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας στην NSA των Ηνωμένων Πολιτειών να υποβληθεί ένα ερωτηματολόγιο με συγκεκριμένες ε, ερωτήσεις προς τον κύριο Σνόουντεν. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό. Ευχαριστώ κύριε Μηγιανμόν, κυρίως που τηρήσατε το χρόνο. Ο κύριος Τονίνο Πίτσουλα. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας συγχαρώ για τα αποτελέσματα που είχατε, ότι ήρθε, ήρθαν δηλαδή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στη Σερβία και Κωσικοπαίδιο. Πριν λυπάμαι για το ότι η κατάσταση στην Ποσνία Ερσεγοβίνη παραμένει ίδια, αλλά βέβαια αυτό είναι αναμενόμενο καθώς υπάρχουν, ε, υπάρχει εσωτερικό αδιέξοδο. Απαιτούνται βεβαίως ε, μεταρρυθμίσεις και πρέπει να δούμε τους πολιτικούς ηγέτες οι οποίοι θα πρέπει να ξεκινήσουν εντατική δουλειά για να έχουν ευρωπαϊκό μέλλον οι πολίτες τους. Ελπίζω πως με το 2013 θα αφήσουμε πίσω μας ε, και την έλλειψη ενδιαφέροντος της διεθνούς κοινότητας για την ε, μοναδική ε, βαλκανική χώρα η οποία δεν έχει πραγματικά ιστορική συνένεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι βλέπετε λοιπόν ε, για το 2014 για την Βοσνία Ζεγοβίνη, καθώς εκεί πέρα θα έχουμε εκλογές και επίσης τι έχετε να πείτε για την μη εφαρμογή της απόφασης του Καστηρίου για τον Φίντσιτ σας ευχαριστώ κύριος ε, Παντσέρη. Θα ήθελα εγώ να κάνω δύο ερωτήσεις. Η, πρώτη, η, από ό,τι κατάλαβα, τα κράτη-μέλη έχουν διάφορες δυσχέρειες. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε λίγο την κατάσταση και τις αμφιβολίες που υπάρχουν για την ε, τάση επεμβάσεων των Γάλλων ε, στην ε, Αφρική. Βεβαίως όλα γίνονται με αποφάσεις του ΙΕ και τα λοιπά, αλλά αυτή η γαλλική παρουσία που έχει λάβει εξοδότηση από την Ευρώπη για να δρά, φαίνεται, αλλά δεν έχει υπάρξει τέτοια εξοδότηση. Είμαστε σε μια περίοδο ε, που δεν είναι πια ε, απικιακή. Είμαστε σε μετα-απικιακή περίοδο, αλλά οι απικιακές δυνάμεις εξακολουθούν να παρεμβαίνουν στις ε, περιοχές των πρώην απικιών τους. Αυτό οπωσδήποτε θα μπορούσε να έχει πολλές παρενέργειες. Δεύτερον, για τη Δυτική Σαχάρα έχω την εντύπωση ότι έχει έρθει πλέον η στιγμή να θέσουμε στην ημερήσια διάταξη το ότι πρέπει εμείς ως, Αφρική, ως Ευρώπη να έχουμε τη δική μας εκτίμηση για το τι συμβαίνει. Συμβαίνει εκεί. Η κυρία Λούψεβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέδι Άστον. Χαίρομαι πολύ για αυτά που μας είπατε και από αυτά που είδα τις ε, ενέργειες της ε, υπηρεσία εξωτερική δράσης. Ευχαριστώ πολύ για αυτά που κάνατε στο Κοσμοπέδιο και τη Σερβία. Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση για τα Βαλκάνια και είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε. Γι' αυτό πιστεύω λοιπόν ότι ε, είστε άξια συγχαρητηρίων. Πρέπει ωστόσο να γίνουν περισσότερε προσπάθειες για την πρώην ε, Ιγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία. Θα πρέπει να γίνουν ε, συζητήσεις και με την Τουρκία, ιδιαίτερα όσον αφορά κάποιες ε, δηλώσεις που κάνει ο Πρωθυπουργός Ερντοάν για βαλκανικές χώρες και οι οποίες ε, προσβάλλονται από τις δηλώσεις αυτές. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι και εδώ υπάρχει ε, απικιακό καθεστώς. Ήταν τμήματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήμουν στη Γεωργία πρόσφατα και σε όλες τις ζητήσεις που κάναμε μας απασχολούσε ιδιαίτερα τους απασχολούσε ιδιαίτερα. Τι θα γίνει ε, στην Ουκρανία, θα υπογράψει η Ουκρανία Συμφωνία Σύνδεσης, θα γίνουν νέες διαπραγματεύσεις, ποια είναι τα κριτήρια που έχουν τεθεί, πόσο εφαρμόζονται. Τώρα για τη Ρωσία. Πιστεύω ότι όπως είπατε και εσείς, οι σχέσεις ε, που έχουμε με τη Ρωσία ε, ε, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πολύ πιο συγκεκριμένα. Θα έχουμε διαπραγματεύσει με τη Ρωσία. Η κυρία Ιάκομ Σάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταία ερώτηση. Εγώ είμαι από το βόρειο της Φιλανδίας, εκεί που ζει ο Άι Βασίλης. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Τι να του πω. Τι θέλετε να ζητήσετε από τον Άι <laughs> Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Να προσπαθήσω να απαντήσω όπως μπορώ. Κύριε Γκαμπριέλ, να ξεκινήσω από εσάς. Η ανησυχία σας ε, για την ε, λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό και την εξαφάνιση των ε, 23 και το ότι πρέπει να αλλάξει πλέον η δομή διαχείρισης ε, κρίσεων ε, πιο μακροπρόθεσμα και να εστιάσουμε και στη διοίκηση και στην ασφάλεια. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε όσον αφορά τις ε, αποστολές ξεκινάμε και δεν ξέρουμε πότε θα φύγουμε, συνεχίζουμε μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις ή να τελειώσουν οι πόροι μας. Και τώρα προσπαθούμε να ορίσουμε μια διάρκεια και ένα στόχο στις αποστολές και βέβαιως προχωράμε κάπως αλλιώς. Αλλά θα δείτε πως ε, τώρα μάλλον πηγαίνουμε από την ε, από την ε, άμεση διαχείριση των ε, κρίσεων και να πάμε κάπως πιο μακροπρόθεσμα και πράγματι θα γίνει νομίζω αυτή η μετάβαση. Ρομπέρτο, σας ευχαριστώ για αυτά τα οποία κάνατε στο Βόρειο Κοσφοπέδιο. Ξέρω πως ε, θεωρείτε πως σας αναζωογόνησε η διαδικασία αυτή. Παίξατε ένα σημαντικό ρόλο στην σύσταση της υπηρεσίας και στην εξέταση, τη σχετική έκθεση και σας ευχαριστώ. Κύριε Σαλαφράγκα, η εξέταση αυτή έγινε ακριβώς για να δούμε τι μπορεί να γίνει βράχη πρόθεσμα, αλλά λέγαμε ουσιαστικά και στα θεσμικά όργανα πως πρέπει να αποφασίσετε κάποια πράγματα να κάνετε. Δεν καλύψαμε τα πάντα και δεν έγινε ε, παρά μόνο για να υπονοήσει πως κάποια πράγματα θα βοηθήσουν στην ε, λειτουργία. Ελπίζω λοιπόν πως ε, θα συνεχιστεί η διαδικασία αυτή. Οπωσδήποτε δεν έχει τελειώσει. Έχουμε βάλει κάποιες βάσεις, αλλά χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Επίσης αυτό το οποίο είπατε για αποσπασμένους ε, εθνικούς εμπειρογνώμονες και έμπειρους ανθρώπους είναι θέμα πόρων το οποίο εγώ θα προτιμούσα να κάνω με τους πόρους τους δικούς μας, αλλά δεν μπορώ γιατί δεν επαρκούν. Οπότε προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τα περιορισμένα κονδύλια που έχουμε σε καιρούς ε, δύσκολους με το καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά επίσης σκεφτόμαστε και όλες τις καταστάσεις που είχαμε τα τελευταία χρόνια, ακόμα και το να ανοίγουμε νέες αντιπροσωπίες όπως έγινε στη Λιβύη, στη Μιανμάρ και θα πρέπει να γίνουμε πιο έξυπνοι στην διαχείριση των κονδυλίων και θα μας βοηθήσετε με κάποιες από τις ε, προτάσεις σας και ξέρω πως θα συνεχίσετε να πιέζετε προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Νταφ, αναφέρατε αρκετά πράγματα. Εγώ θα αναφερθώ ειδικά στις ε, μονάδες ε, μάχης και τον σκοπό που έχουν. Ξέρετε, είναι πολύ ενδιαφέρον να κοιτάμε τα διάφορα μέσα, όπως τα λέμε, και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά. Όσον αφορά την αποστολή της Γαλλίας, είμαστε σε στενή επαφή με την Γαλλία. Είναι μια αποστολή που ξεκίνησε η Γαλλία μόνη της. Δεν έχει σχέση με απεικιοκρατία. Είναι θέμα ιστορικών δεσμών και στήριξης ε, της χώρας ε, στο μέλλον. Ε, αλλά βεβαίως προσπαθούμε να βρούμε στήριξη και από άλλες χώρες και οπωσδήποτε ο κύριος Ολάντ θα το αναφέρει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ένα ζήτημα πολύ δύσκολο είναι πώς μια διαδικασία λήψη αποφάσεων με 28 συμμετέχοντες να μπορεί να κινηθεί γρήγορα. Για διάφορους λόγους. Όταν ε, συναντώνται άνθρωποι από διαφορετικές ε, χώρες ε, και πρέπει από κοινού να εκτελέσουν μια αποστολή, ε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Κανόνες εμπλοκής, το τι πρέπει να κάνουν, σχεδιασμός. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό με ταχύτητα που θα θέλαμε ακόμα. Αλλά βεβαίως ε, σημαντικό είναι οι πολιτικές αποφάσεις ε, να λαμβάνονται από τις χώρες που θα στείλουν τους ανθρώπους τους. Να κινδυνεύσουν έτσι. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε πως πρέπει να λειτουργεί αυτό το δίκτυο με τρόπο συνενετικό. Υπό αυτές τις συνθήκες νομίζω πως η προσέγγιση της Γαλλίας, δηλαδή να μπει και ε, να, δει, να δώσει δηλαδή μερή βοήθεια και να μιλήσει μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δει το τι μπορεί να γίνει για τη στήριξη της αποστολής και βεβαίως γιατί στο Μαλί υπάρχει αποστολή η εκπαιδευτική και η μακροπρόθεσμη αποστολή αναπτυξιακή νομίζω πως είναι ένα καλό παράδειγμα του τι μπορούμε να κάνουμε και εξετάσαμε όλες μας τις επιλογές. Κύριε Σούλτς, με ρωτήσατε για το εάν η Ουκρανία θα αναγκαστεί να μην έχει πλέον τέτοια σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, δεν νομίζω και ελπίζω ειλικρινά να μην συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά πραγματικά πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά το τι γίνεται με την ανατολική μας ε, εταιρική σχέση, να μπορούν οι χώρες να λαμβάνουν τις αποφάσεις που θέλουν και να τις στηρίζουμε και προσφερθήκαμε προσφέραμε τις υπηρεσίες μας για οποιαδήποτε μεσολάβηση. Μίλησα με τον πρόεδρο, εκείνος ζήτησε τη δική μου συμμετοχή. Εγώ είπα ευχαρίστως εάν παίξει αυτό κάποιο ρόλο. Αλλά πρέπει να ξέρουμε και ποιος είναι ο ρόλος ο οποίος μας προτείνεται. Εγώ όταν μίλησα με τους ηγέτες της αντιπολιτευσής είπα πως μπορούμε να εμπλακούμε με διάφορους τρόπους. Έχουμε παίξει διάφορους ρόλους. Ε, του διαπραγματευτή, του διαμεσολαβητή. Και εγώ που ταξιδεύω κάθε φορά ανά την Ιφίλιο, παίζω διαφορετικό ρόλο κάθε φορά, αλλά δεν τίθεται ζήτημα πως υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι σε θέση και θέλουν να στηρίξουν ε, την διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην δική μας την υπηρεσία, αλλού και βεβαίως έχουμε κάθε διάθεση. Οπότε, αν θελήσουν κάτι τέτοιο οι Ουκρανοί, είμαστε στην διάθεσή τους, αλλά πρέπει να το θέλουν. Και Στυρ με ρωτήσατε για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Ναι. Έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά στην Βοσνία Ζεγοβίνη. Είχα μία συζήτηση τεσσάρων ωρών για το ακριβώς τι πρέπει να γίνει από εδώ και μπρος πριν από λίγες ημέρες. Ο Στέφεν έκανε πολύ καλή δουλειά όσον αφορά το να συνομιλήσουν οι διάφοροι ηγέτες, αλλά πρέπει να δούμε ξανά το πώς θα στηρίξουμε αυτή τη χώρα, η οποία κινδυνεύει να μείνει πίσω ε, στην περιοχή και επίσης πώς θα χρησιμοποιήσουμε την πύρα που υπάρχει στην περιοχή. κυβερνήσεις που έρχονται πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιτυχία με τη Σερβία και το Κοσμοπέδιο που όλοι έλεγαν πως δεν έχει καμία πιθανότητα. Πώς θα αναπτύξουμε λοιπόν από εδώ και μπρος μια στρατηγική για την Βοσνία Ζεγοβίνη για το μέλλον. Φαίνεται να έχει κολλήσει η υπόθεση. Οπότε συμφωνώ μαζί σας. Πρέπει να σκεφτούμε πράγματι τους μοχλούς πίεσης ε, που υπάρχουν και στην περιοχή. Αλλά όπως σας είπα το θέμα είναι ολόκληρα τα Δυτικά Βαλκάνια να έρθουν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οπωσδήποτε θα μας απασχολήσουν του χρόνου. Γιατί θέλω πράγματι ο κόσμος να τα πάει καλύτερα. Βερονίκα, ευχαριστώ για την επιστολή σας. Θαυμάσια. Θα παίξουμε νομίζω σημαντικό ρόλο στην, στο δεύτερο κύριο της για διάφορους λόγους. Πρώτον, εμείς εδώ και δύο χρόνια λέμε πως πρέπει να υπάρχει μια πολιτική διαδικασία. Εμείς υποστηρίζαμε τον πρώτο γύρο της Γενέβης, ο Πιέρ Δημόν, όπως είπα, συναντάει τους ε, τα μέρη. Ο κύριος Μπραχήμη επίσης ε, προετοιμάζει τον δεύτερο γύρο και πάλι θα συναντηθούν κάποιοι στη Γενέβη για να στηρίξουν την προσπάθεια του ΟΗΕ. Οπωσδήποτε παίζουμε ένα ρόλο κλειδί για να εμπλακεί και η κοινωνία των πολιτών και πιέζουμε, όπως είπα, οι γυναίκες να βρίσκονται σε κάθε αντιπροσωπεία. Πρέπει να πω πως ο ΙΕ πάντα λέει στις αντιπροσωπείες πως αναμένει να έχουν και οι γυναίκες ως μέλη. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό. Και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα από εδώ και μπρος για να αναγνωριστεί ότι είμαστε και οι μεγαλύτεροι δωρητέ ε, και υποστηρικτέ όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια. Θα παίξουμε λοιπόν αυτό το ρόλο και θα είναι πολύ σημαντικό. είναι πολύ σημαντικό να είμαστε σε επαφή με όλου για να υπάρχει επιτυχία. Για τον Νότιο Σουδάν. Είναι δύσκολο να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει λόγω των όσων συμβαίνουν με την ομάδα αυτή, το SPLM. Όπως είπα, Υπάρχει, ε, εξελίσσεται αυτή τη στιγμή μια συνάντηση στην οποία δεν βρίσκομαι. Το αεροδρόμιο έχει κλείσει, ο εναέριος χώρος ε, επίσης. Οπότε προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε πρώτα απ' όλα αυτούς που βρίσκονται εκεί πέρα για ανθρωπιστική εργασία. Ε, τώρα δεν ξέρουμε τι γίνεται, αν είναι σποραδικές οι συγκρούσεις, αν έχει ξεφύγει η κατάσταση εκτός ελέγχου, εκτός της ε, Τζούμπα. Ε, επίσης είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο Εξωτερικών της Αιθιοπίας που είναι σε επαφή με τον Νότιο Σουδάν και αναμένουμε νεότερες πληροφορίες. Περίμενα εδώ πέρα νέες πληροφορίες, αλλά κάθε φορά ε, οι πληροφορίες είναι αντιφατικές, οπότε πρέπει να έχουμε κάποια πράγματα πιο σίγουρα. Αλλά όπως είπατε έχουμε μια αποστολή εκεί πέρα που κάνει καλή δουλειά, αντιπροσωπεία. Όλοι είναι ασφαλείς. Πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει ηρεμία και βεβαίως ε, και ο πρόεδρος νομίζω προσπαθεί να ηρεμήσει την κατάσταση. Κύριε Βίγκελ, αναφερθήκατε στην Ουκρανία και τις διαφορές μεταξύ της Ανατολικής και της Δυτικής Ουκρανίας. Ορισμένοι λένε ότι είναι περίπου δύο χωριστές χώρες. Όχι, εγώ δεν θα το περιέγραφα έτσι. Νομίζω ότι είναι μια χώρα που αναπόφευκτα έχει ε, έντονους δεσμούς με δύο ε, κατευθύνσεις. Για πολλές ε, εταιρείε στην Ανατολική Ουκρανία η κύρια αγορά τους είναι η Ρωσία και θα παραμείνει. Και είναι φυσιολογικό. Άλλα τμήματα της χώρας κοιτάνε προς αλλού, προς τα σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό όταν, προσπαθούμε να... όταν προσπαθούν να διαμορφώσουν την πολιτική τους, να το σκεφτούν σωστά. Δηλαδή αυτά που προτείνουμε εμείς να μην εμποδίσει τη συνέχιση της ε, πολύ εκτεταμένης ε, συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου και οικονομικών δεσμών με τη Ρωσία. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει λοιπόν η στρατηγική μας να αφορά όλη την Ουκρανία, να μην προσπαθούμε να διχάσουμε τη χώρα. Κύριε Μιλιάν, με ρωτήσατε τι είπαμε στο γεύμα με τον Σαργέη Λαμπρόφ. Πολύ ενδιαφέρον γεύμα. Α το πω έτσι. Κοιτάξτε, σε αυτές τι περιπτώσει δύο προσπαθούμε να επιτύχουμε. Πρώτον, να μιλήσουμε για την ε, επερχόμενη συνάντηση κορυφής του Ιανουαρίου και το ενδεχόμενο στρατηγικού διαλόγου για την ανάπτυξη σχέσεων με τη Ρωσία και τα διμερεί θέματα που μας απασχολούν. Υπάρχει σημαντική κινητικότητα για αυτή τη νέα συμφωνία. Ελπίζουμε ε, Αυτά αποτελέσματα για να αρχίσουμε να συζητάμε και την πλευρά εμπορίου και επενδύσεων. Αυτό εξετάζουμε τώρα. Ελπίζω τις επόμενες εβδομάδες να έχουμε αποτελέσματα. Αλλά είναι σαφές ότι η Ρωσία θέλει επίσης να έχει στενούς δεσμούς με τους γειτονές της. Και για τον πρόεδρο Κούπιν, Πούτιν η Τελωνιακή Ένωση είναι σημαντική πολιτική και οικονομική προσπάθεια και οι σχέσεις ε, της Ρωσίας με τους ανατολικούς της εταίρους, με τους δυτικούς της εταίρους, με τους οποίους εμείς έχουμε επίση σχέσεις, είναι σαφές ότι είναι σημαντικό, γιατί οι χώρες αυτές βέβαια δεν επιδιώκουν το ένα ή το άλλο, θέλουν και τα δύο. Είναι λογικό και εμείς ε, αναμένουμε να έχουν ε, στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, αλλά και εμείς θα θέλαμε να έχουμε ωφέλη από τη δική μας καλή σχέση με αυτούς. Με ρωτήσατε για την απόφασή σα να καλέσετε τον κύριο Σνόντεν. Αυτό είναι δικό σα θέμα, δεν με αφορά. Δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Εμεί συνεργαζόμαστε, να, συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ για το θέμα του NSA. Μίλησα με το Σύμβουλο Ασφαλεία, το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας και το καθιστούμε πάντα σαφέ. Θα ακούσατε και διάφορε ενημερώσει για τη δουλειά που κάνει η κυρία Ρέντινγκ και άλλοι για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτά τα θέματα. Κύριε Πεκούλα, αναφερθήκατε στην ε, Βοσνία Ζεγοβίνη. Χαίρομαι που επανέρχεται στο προσκήνιο. Συζήτησα επί μακρόν για να καταλάβουν οι συνάδελφοι και στα κράτη-μέλη και στις υπηρεσίες και στην Κομισιόν πώς πρέπει να προωθήσουμε το θέμα αυτό. Πώς θα καταδείξουμε ότι το μέλλον αυτής της χώρας ε, είναι πολύ στενά συνδεδεμένο με την Ένωση, ότι όλη η περιοχή οδεύει προς την Ένωση. Υπάρχουν πολλοί ενδιαφέρουσες ευκαιρίες, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουν μερικά από τα ε, θέματα. Η συγκεκριμένη απόφαση του δικαστηρίου είναι ένα τμήμα, αλλά όχι μόνο. Και επίσης να υπάρξουν ε, αποφασιστικοί πολιτικοί ηγέτες σε όλα τα τμήματα της Βοσνίας της που να αρχίσουν να συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν και τις οικονομικές προκλήσεις αλλά και μερικά πολιτικά θέματα. Είναι λοιπόν ένα θέμα που ελπίζω να επανέλθουμε και ελπίζω να σημειωθεί πρόοδος. Κύριε Παντζέρη, όπως είπα και προηγουμένως, η γαλλική συμμετοχή στην κεντροαφρικανική δημοκρατία είναι ιστορικό θέμα. Θέσατε το θέμα της Δυτικής Σαχάρας. Συνεργαζόμαστε, όπως πάντα, με τα Ηνωμένα Έθνη για το θέμα αυτό και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Πολλά θέματα, ωστόσο, που αντιμετωπίζουμε με πολλές χώρες, σχετίζονται με τους ιστορικούς ε, δεσμούς ή τις μακροχρόνιες συμφωνίες που έχουν ε, κάποιες κάποια κράτη-μέλη με αυτές τις περιοχές. Αυτό σημαίνει επίσης ότι στο Συμβούλιο έχουμε πολύ γνώση και εμπειρία. Άλλοι έχουν στενή σχέση με την Λατινική Αμερική, άλλοι με τμήματα της Αφρικής και της Ασίας. Έχουν ιστορία κοινή, πείρα, δεσμούς, οπότε αυτό εμπλουτίζει την εργασία της υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Κύριε Διόψεβα, με ρωτήσατε μια σειρά θέματα, αλλά ο ρόλος της Τουρκίας ε, για τα Δυτικά Βαλκάνια. Να μιλήσω γι' αυτό. Και μετά θα μιλήσω και για Ρωσία-Ουκρανία. Η Τουρκία είναι πολύ σημαντικό εταίρο για πολλά θέματα που κάνουμε στην εξωτερική πολιτική, για πολλά θέματα γειτονία. Και πολλέ συζητήσει για την Βοσνία-Ερζεγοβίνη στρέφονται γύρω από τον σημαντικό ρόλο των σχέσεων της Τουρκίας με τα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία ενεργά συνεργάζεται μαζί μας για να υποστηρίξει την πορεία των Δυτικών Βαλκανίων προς την Ένωση. Και επίση έχουν βοηθήσει στις σχέσεις μας με το Ιράν. Στις σχέσεις μας με το Ιράν. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το τμήμα της συζήτησης. Δηλαδή μας βοηθούν οι Τούρκοι ε, σε πολλά θέματα όπως και άλλες χώρες μας βοηθούν σε άλλα θέματα. Λοιπόν, τι να μου φέρει ο Άι Βασίλης. Θα ήθελα ε, ε, πολλοί λαοί και ιδίω ο λαό τη Συρία να περάσουν καλύτερα Χριστούγεννα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία εκπρόσωπε. Η κυρία Γκόμες. Κυρία Κρίσμας, έρχονται τα Χριστούγεννα. Και είπατε ότι ο κύριος Μπαρόζο ε, συνομιλεί με την Αιθιοπία. Μπορείτε να του ζητήσετε την απελευθέρωση των, ε, εθοποιών, των ε, πολιτικών κρατουμένων της Αιθιοπίας όπως η κυρία Ρία Λέμο η οποία είναι φυλακισμένη ενώ υποφέρει από καρκίνο ε, του μαστού και δεν έχει καμία θεραπεία στη φυλακή όπως μας είπε η αδελφή της με την οποία πρόσφατα μιλήσαμε. Υπάρχει άλλο αίτημα. Ευχαριστώ Λέδη Άστον για την δράση σας, τη δέσμευσή σας, για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ.